Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ελπίζω ότι περάσατε όμορφες καλοκαιρινές διακοπές και ότι η καινούργια αυτή περίοδος θα είναι μια σημαντική χρονική περίοδος για την Επιτροπή μα Επιτροπή ανάπτυξη και ότι θα πετύχουμε σημαντικούς στόχους, ιδιαίτερα όσον αφορά την καταπολέμηση των αλλαγών του κλίματος και ότι θα δουλέψουμε υπέρ των υποανάπτυξη χωρών. Ξεκινάμε εγκρίνοντας την ημερήσια διάταξη. Υπάρχουν αντιρρήσεις, παρακαλώ, ή σχόλια για αυτό το σχέδιο ημερήσια διάταξης που έχετε μπροστά σας. Όχι από ό,τι βλέπω, οπότε εγκρίνεται. Έχουμε πρακτικά τώρα των προηγούμενων συνεδριάσεών μας. Η 21η-22η Ιουνίου 2010, 1η Ιουλίου 2010 και 5η Ιουλίου 2010. Τα έχετε πάρει όλοι. Αν τυχόν έχετε παρατηρήσεις επί των πρακτικών αυτών, παρακαλώ να το πείτε στη γραμματεία πριν τη λήξη της ε, συνεδρίασής μας. Αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα. Τώρα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μια έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής μας θα λάβει χώρα αύριο. 2 με 3,5 στην αίθουσα 5G2 και θα αφιερωθεί στις καταστροφικές πλημμύρες που είχαμε στο Πακιστάν και στην τεράστια ανθρωπιστική κρίση που προκάλεσαν οι πλημμύρες αυτές. Η Ερμόδια επίτροπος για την ανθρωπιστική βοήθεια, η Κρυσταλίνα Τσάτσεβα, θα έρθει, η Κρυσταλίνα Τζόρτζεβα λοιπόν, θα έρθει για να μας μιλήσει για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση αυτή και να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή της επιτόπου. Πήγε εκεί 23 με 25 Αυγούστου. Συνεπώς, βασίζομαι σε εσά, την παρουσία σας, για την τόσο σημαντική αυτή συνεδρίαση που μας υπαγορεύει η επικαιρότητα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να ανακοινώσει κάτι, μήπως? Όχι, από ό,τι βλέπω. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε λάβει προς το παρόν καμία ερώτηση που να απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν έχουμε ερωτήσει σήμερα. Και τώρα περνάμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι η εφαρμογή ορισμένων κατευθυντηρίων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που την χάνουν δημόσιας στήριξης. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που δεν είναι τόσο γνωστό αλλά πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των χωρών του Νότου. Η αλήθεια είναι ότι οι παρατηρητέ ε, συζητούν τα υπέρ και τα κατά των εξαγωγικών αυτών πιστώσεων. Οι δραστηριότητε των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων θεωρούνται από ορισμένου σαν κάτι θετικό για την ανάπτυξη μεγάλων εταιριών και επιχειρήσεων, αλλά άλλοι επικρίνουν τους οργανισμούς αυτούς διότι φοβούνται ότι εκεί που γίνονται οι επενδύσεις γίνονται σε βάρος πολιτικών που είναι ε, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων των μισθωτών. Η των δικαιωματων των μισθωτων η συγκητη μας για γνωμοδότηση είναι ο Μπάρτ Στάς. Η γνωμοδότησή του απευθύνεται στην Επιτροπή ΙΝΤΑ που είναι και αρμόδια επί της ουσίας για την απόφαση που θα πάρει το Συμβούλιο όσον αφορά κατευθυντήριες γραμμές για τις εξαγωγικές πιστώσεις που έχουν ε, δημόσια στήριξη. Πρόκειται Βέβαια, για το πώς θα συμπεριλάβουμε τη διάσταση της ανάπτυξης της κατευθυντήρησης σε αυτές γραμμές, ώστε οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων να λαμβάνουν υπόψη τις αρχές μας και τον αγώνα μας για την καταπολέμηση της ένδειας και προκειμένου οι πολιτικές μας και οι πολιτικές των οργανισμών αυτών να συνάδουν με τους στόχους της ανάπτυξης. Έχουμε ένα έγγραφο εργασίας που το έχετε πάρει όλοι. Οπότε πάνω σε αυτό θα συζητήσουμε. Κύριε Στάση, έχετε το λόγο λοιπόν για έξι λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ακούγεται πολύ τεχνικό το θέμα αυτό, όμως ε, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και είναι πολύ σημαντική η γνωμοδότηση που ετοιμάζουμε εμείς ε, για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Οι οργανισμοί εξαγωγικών ε, ε, για εξαγωγές και επενδύσεις είναι ένας οργανισμός πολύ σημαντικός και στόχος του έχει να χρησιμοποιεί χρήματα των φορολογούμενων για να κάνει λιγότερο αβέβαιες τις εξαγωγές και τις επενδύσεις στο εξωτερικό εκ μέρους των τοπικών επιχειρήσεων. θέλουμε ακριβώς να αποφύγουμε τις αβεβαιότητες που υπάρχουν, που δύσκολα ασφαλίζονται. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα διαφόρων οργανισμών που φροντίζουν για εξαγωγικές πιστώσεις, στον ιδιωτικό τομέα για παράδειγμα. Άλλοι πάλι στηρίζονται από το κράτος και άλλοι είναι καθαρά κυβερνητικοί οργανισμοί. Οι συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν καλά τα τεχνικά στοιχεία θα έχουν αν μη τι άλλο ακούσει κάποιους τέτοιους οργανισμούς. Για τη Γαλλία έχουμε την ΚΟΦΑΣΕ για την ε, Ολλανδία η Radius. η Φινβέρα στη Φιλανδία, στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι η Export Credit Guarantee Portmans, στη Γερμανία έχουν την Euler Hermes. Τώρα οι κανόνες που ισχύουν για τις εξαγωγικές πιστώσεις για τις χώρες ΟΣΑ ε, βασίζονται σε κάποιες συμφωνίες που έχουν γίνει. Μέσα στον ΟΣΑ που όμως δεν είναι δεσμευτικές. Πλαισιώνουν όμως το θέμα αυτό και έτσι καλύπτονται οι κυβερνήσεις που προσφέρουν αυτές τις εξαγωγικές πιστώσεις. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθήσαμε να ετοιμάσουμε ένα policy paper από τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες που ισχύουν. Πάντως, το στοιχείο κλειδί στην όλη υπόθεση είναι η συμφωνία στον ΟΣΑ, που είναι η διαρρύθμιση που γίνεται από την ομάδα εξαγωγικής πίστοσης και που λέει ότι ε, το κείμενο αυτό του ΟΣΑ, η συμφωνία αυτή του ΟΣΑ πρέπει να γίνει και κείμενο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάσει της συνθήκης της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποκτά περισσότερες αρμοδιότητες για αυτό το θέμα. Δηλαδή η συνθήκη τη Λισαβόνα λέει ότι αυτά τα οποία συζητάμε βάσει τη ε, συνήθους νομοθετική διαδικασία από το Κοινοβούλιο, από την Επιτροπή μας, έχει μεγαλύτερο βάρος και επιρροή. Και γι' αυτό εμείς πρέπει να φροντίσουμε τι κατευθυντήριε γραμμέ που έχουμε από τον ΩΣΑ να τι κάνουμε ευρωπαϊκή νομοθεσία αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή ΙΝΤΑ. Εμείς πρέπει να γνωμοδοτήσουμε έτσι ώστε να υπάρξει και διάσταση της ανάπτυξης στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές. Γιατί τώρα θέλουμε ή θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές να γίνουν Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό είναι για να είμαστε περισσότερο σίγουροι όσον αφορά τις εξαγωγικές αυτές πιστώσεις, ότι δηλαδή δεν θα βοηθούν αμφιλεγόμενα προγράμματα, ούτε θα ακολουθούν μηχανισμούς αμφιλεγόμενους υπέρ του διεθνούς εμπορίου. Αν διαβάσετε τόσο έχουν γραφεί αυτό το θέμα, θα δείτε ότι το θέμα των εξαγωγικών πιστώσεων και των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλές ερωτήσεις. Κατά πώς υπάρχει αρκετή διαφάνεια, κατά πώς υπάρχει αρκετός έλεγχος κατά πόσο υπάρχουν εγγυήσει ότι διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι καταπολεμείται η διαφθορά, ότι δεν ε, ερχόμαστε εδώ σε αντίφαση με άλλους στόχους που είναι υπέρ του περιβάλλοντος, για παράδειγμα. Η χρηματοδότηση ε, ε, επίσης που δίνει κάθε οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων οδηγεί μερικέ φορέ αφιλεγόμενα έργα. Για παράδειγμα, στη δικιά μου χώρα επρόκειτο για εξαγωγέ όπλων που χρηματοδοτήθηκαν από εκεί. Όπω επίση διάφορα προγράμματα υποδομών που είναι αφιλεγόμενα. Και μάλιστα μερικές φορές έχουν χρηματοδοτηθεί και έργα τα οποία αρχικά είχαν απορριφθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ως λοιπόν Επιτροπή Ανάπτυξης θέλουμε να εξετάσουμε την προβληματική αυτή των εξαγωγικών πιστώσεων ώστε να φροντίσουμε να μην συμβαίνει αυτό πια, να μην είναι αμφιλεγόμενα δηλαδή τα έργα, να υπάρχει διαφάνεια, να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Να υπάρχει ασφάλεια δικαίου παραπάνω για τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Μην ξεχνάμε και τους στόχους της χιλιετίας. Δεν θέλουμε και αυτοί να πάνε πίσω εξαιτία τέτοια χρηματοδότησης. Συχνά οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων δίνουν ε, τα χρήματά τους μέσω του κλαπ του Παρισιού. Πρόκειται για μια συμφωνία κοινών προσεγγίσεων που έχει όμως πολλές ασάφειες. Οι χώρες οι οποίες παίρνουν τα χρήματα, διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές ε, τα χρήματα αυτά επηρεάζουν την αναπτυξιακή βοήθεια. Και γίνεται ένα μπέρδεμα για ανάμεσα στην αναπτυξιακή βοήθεια και τις εξαγωγικές πιστώσεις. Οι χώρα ΩΣΑ επίσης πολλές φορές αυτό που κάνουν είναι ότι τα χρεολύσια για ε, τις πιστώσεις αυτές τις συμπεριλαμβάνουν στατιστικά σε άλλες ομάδες, κάτι το οποίο μπερδεύει βέβαια πολύ τα πράγματα. Στο έγγραφο εργασίας μου θα δείτε ότι αναφέρονται διάφορα σημεία απαριθμημένα για το τι προτείνει ο εισηγητής σας προκειμένου να τροποποιηθεί η πρόταση και να συμπεριληφθούν τα σημεία αυτά στη νέα νομοθετική πρόταση. Για παράδειγμα, θέλουμε η συμφωνία του ΟΣΑ που θα γίνει νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι πλήρως συμβατό αυτό με τους στόχους του άρθρου 208 της συνθήκης που έχει να κάνει με την δημοκρατία, με το κράτος δικαίου, το σεβασμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιώδες ελευθερίες κλπ. Επίσης, οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό πρέπει αυτό να το κάνουν μόνο εφόσον οι εξαγωγικές πιστώσεις που δέχονται κρατική στήριξη δεν επηρεάζουν αρνητικά τις αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση, για παράδειγμα, με την εκπλήρωση προηγούμενων διεθνών, περιφερειακών ή εθνικών υποχρεώσεων που έχουν, είτε πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, είτε πρόκειται για την κοινωνική πολιτική, είτε για το περιβάλλον. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε ότι εφόσον υπάρχει κάποια χρηματοδότηση να μην πλήττεται η στρατηγική των χωρών ε, αυτών ε, στο πλαίσιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ή άλλων αρμοδίων διεθνών οργανισμών. Επίσης, πρέπει να υπάρχει ανεξάρτητος έλεγχος, τακτικά. Και να βγαίνει προς τα έξω δημόσια μια έκθεση που να βασίζεται σε έλεγχο ώστε οι δραστηριότητες αυτές των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων να συμβάλλουν στο γενικό στόχο της Ένωσης που αναφέρεται στο άρθρο 28 της Ειδικής της Λισαβόνας. Επίσης κάτι το οποίο ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ στην Προεδρό μας, ότι οι κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι τέτοιε, ώστε όλες οι διεθνεί συμβάσει και οι συνθήκες να τηρούνται εκείνες δηλαδή που αναφέρονται στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Το ίδιο και για μελέτες περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Να γίνονται τέτοιες μελέτες πριν υπάρξει χρηματοδότηση. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουν οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων να έχουν λεπτομερείς πολιτικές προσφοράς πληροφοριών. Κάτι άλλο για το οποίο έχουμε συχνά μιλήσει εδώ στην Επιτροπή μας είναι οι κλιματικές αλλαγές. Ε, λοιπόν, οι νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές πρέπει να είναι έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Το σημείο 7 λέει ότι πρέπει να σταματήσει να καταγράφεται η αποπληρωμή εξαγωγικών πιστώσεων ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και τέλος, με κάποια τροπολογία πρέπει να φροντίσουμε να λέμε ότι ό,τι χρέη έχουν δημιουργηθεί, το οποίο όμως δεν ε, καλύπτουν τις απαιτήσει διαφάνειας ή ως προς το νομικό χαρακτήρα, δεν καλύπτουν κοινωνικές και προδιαγραφές, να ακυρωθούν τα χρέη αυτά. Σας είπα λοιπόν ποια είναι η άποψή μου. Με τον εισηγητή από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου έχω συμφωνήσει ότι θα βρεθούμε για να συζητήσουμε τις τροπολογίες αυτές που προτείνω. Στα τέλη αυτού του μήνα θα είμαι έτοιμος πιστεύω. Αρχές Οκτωβρίου θα μπορέσουμε να συζητήσουμε την έκθεση εδώ στην Επιτροπή αυτή Ανάπτυξης. Μετά θα ξεκινήσει η περίοδος για την κατάθεση τροπολογιών. Συνεπώς, μέσα Οκτωβρίου θα μπορέσω, φαντάζομαι, να έχω προσαρμόσει την έκθεσή μου βάσει των τροπολογιών που θα προτείνετε, να την εγκρίνουμε και τον Δεκέμβριο να φτάσει στην Ολομέλεια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής πάντως πρέπει να ξέρετε ότι είχα συχνά επαφές και με τον εισηγητή από την Ίντα αλλά και με την Βελγική Προεδρία. Γιατί είναι σημαντικό να προχωρήσει αυτή η υπόθεση κατά τη διάρκεια της Βελγικής ε, Προεδρίας. Καλό θα ήταν λοιπόν να προχωρήσουμε ε, χέρι-χέρι με το Συμβούλιο για να καταλήξουμε σε αυτήν την ε, νομοθετική απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τόσο σημαντική σας δουλειά που μοιραστήκατε μαζί μας. Τώρα το λόγο έχουν οι ευρωβουλευτές. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο παρακαλώ. Εγώ έχω να κάνω ένα μικρό σχόλιο, επιτρέψτε μου. Πιστεύω ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις, εφόσον είναι καλά ρυθμισμένες, είναι πολύ καλές για να καταπολεμάμε ακριβώς την διαφθορά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπεί ο κύριος Ντενίρε Ντονέ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ε, θέλω μόνο να πω ότι εξετάσαμε πολύ προσεκτικά το έγγραφο εργασία ε, του εισηγητή σα. Ήδη ε, συνεργαζόμασταν στενά με τον εισηγητή τη ΙΝΤΑ ε, και από πλευρά τη Επιτροπή ω θέμα αρχή καλωσορίζουμε την έμφαση που δίδεται στο έγγραφο αυτό καθώ και στη συζήτηση που μόλι είχαμε στην Επιτροπή την έμφαση που δίνεται λοιπόν στη διαφάνεια στο επίπεδο της Ένωσης όσον αφορά τον τομέα πολιτικής των εξωτερικών πιστώσεων και το έλεγχο στον οποίο, τον οποίο θα ασκήσει το Κοινοβούλιο σε αυτήν τον τομέα πολιτικής όπως και σε τους υπόλοιπους και βεβαίως εμείς από πλευρά της Κομισιόν θα μεριμνήσουμε, θα φροντίσουμε να διατηρηθεί η αρχική λογική της πρότασής μας που σημαίνει την μεταγραφή του διεθνούς, ε, μάλλον στο κοινοτικό νομοθεσία, της διεθνούς νομοθεσίας, μεταγραφή στο κοινοτικό, στην κοινοτική, κοινοτική νομοθεσία των προσεγγίσεων του ΟΣΑ, τις άλλες ε, προδιαγραφές που υπάρχουν φυσικά στο πλαίσιο του ΟΣΑ, αλλά και για άλλα μέσα ισχύουν αυτές οι ίδιες προδιαγραφές. Αν λοιπόν αυτό είναι ο προσανατολισμός του Κοινοβουλίου, θα εμπλακούμε και εμείς σε αυτή τη συνεργασία, σε οποιαδήποτε πρόταση ε, έτσι ώστε ε, να βελτιωθεί όσο γίνεται η διαφάνεια με την προϋπόθεση ότι τέτοιες ε, διατάξεις θα είναι δυνατόν να ε, επιβληθούν ε, από τεχνικής άποψης, ότι δεν θα έρχονται σε σύγκρουση με τις υφιστάμενες διατάξεις περί διαφάνειας σε επίπεδο ένωσης αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Και τέλος, κυρία Πρόεδρε, διατάξεις ή προτάσεις για περαιτέρω απαιτήσει διαφάνειας θα συμφωνήσουμε στο βαθμό που δεν επιβαρύνουν τις τρίτες χώρες και τις δικές μας δυνατότητες ε, προσφοράς στήριξης στους Ευρωπαίους ε, εξαγωγείς με βάση βέβαια τις αρχές του ΠΟΕ. Πράγμα το οποίο είναι και η βασική μέρημνα αυτής της πρότασης της Κομισιόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό το θέμα τον Οκτώβριο. Προχωράμε τώρα στο σημείο 7, Διεθνής Εμπορική Πολιτική, στο πλαίσιο των επιταγών ε, των κλιματικών αλλαγών. Η συνάδελφος Κατερίνα Γκρέσλε μας παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησης επί της ε, Έκθεση που έχει συνταχθεί στην ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ σε σχέση με τη διεθνή πολιτική στο πλαίσιο των επιταγών της αλλαγής ε, του κλίματος. Συνοχή λοιπόν της πολιτικής ε, περιβάλλοντος, επαλήθευση του συνόλου των πολιτικών της Επιτροπής, της ε, Ένωσης μάλλον, ότι δηλαδή προχωρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Γκρέζ, έχετε έξι λεπτά για να μας παρουσιάσετε ε, την έκθεσή σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Αυτό το θέμα της ε, ένταξης της κλιματικής πολιτικής, της εμπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι εξαιρετικά σημαντικό και είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας εδώ, στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Η κρίση μας έδειξε πως χρειάζεται περισσότερες ρυθμίσεις, περισσότερη συνεργασία, ώστε να διατηρηθεί αυτό που καλείται το, τα, τα δημόσια αγαθά, το κλίμα, το νερό, η βιοπικιλότητα. Η κρίση μας έδειξε επίσης ότι οι κλιματικές αλλαγές και ακριβώς αυτό το τομέα ε, μπλέκεται ιδιαίτερα η Επιτροπή Ανάπτυξης, ε, πλήττει κυρίως ε, τις ε, χώρες που είναι υπό ανάπτυξη. Βλέπουμε λοιπόν ήδη 300.000 ε, νεκρούς. Δεν πρόκειται για λούξια πολυτέλεια, αλλά για κάτι το απόλυτα απαραίτητο, το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Να θυμίσω τα ενένεια των Ηνωμένων Εθνών για διαφοροποιημένη κοινή ευθύνη, που σημαίνει ανάληψη ευθύνης από πλευρά των πιο αναπτυγμένων χωρών, ιδιαίτερα όσον αφορά την προσαρμογή της εμπορική τους πολιτικής. Και αυτό, και αυτό το είδαμε κατά τη διάρκεια των εργασιών μας, ε, καθώς επιπλέον τα πήγοντα μέτρα τα οποία λαμβάνονται για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, συχνά δεν αφορούν την βοήθεια για την ανάπτυξη και αυτό είναι το οποίο εμείς ε, θα θέλαμε. Το καλό είναι ότι θα πρέπει να είναι αρκετά εύκολα τα πράγματα και να μπορούν να ενταχθούν όλες αυτές οι κλιματικές, ε, μάλλον οι πολιτικές ανάπτυξης μέσα στην εμπορική πολιτική. 20% των εκπομπών ε, αερίων του θερμοκηπίου οφείλονται στην ε, παραγωγή ενέργειας. Είναι προφανές ότι η παραγωγή ενέργειας θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τις μεθόδους που καταναλώνουν λιγότερο, μάλλον που εκπέμπουν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα. Υπάρχει μια σχετική ανάπτυξη εδώ. Ένα δεύτερο σημείο και είναι ένα καλό παράδειγμα για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει η πολιτική μας σε θέματα γεωργίας. Δηλαδή και εκεί γνωρίζουμε πολύ καλά πως μια γεωργία που είναι ταυτόχρονα βιολογική αλλά και με μικρά κυκλώματα ε, δημιουργεί λιγότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Ε, τρίτο σημείο είναι η αγορά άνθρακα. Εδώ το έχουμε ήδη εξετάσει το θέμα, το γνωρίζουμε όλοι αυτό. Λειτουργεί άσχημα. Οι μηχανισμοί ίδια ανάπτυξη έχουν ήδη αποδείξει ότι είναι ανεπαρκείς, ότι δεν λειτουργούν σωστά. Και τέλος, δεν θα ξεφύγουμε από την ε, θέσπιση μιας, ε, ενός φόρου για προϊόντα τα οποία ενσωματώνουν ε, την περιβαλλοντική διάσταση. Τέταρτο σημείο το οποίο θα ήθελα να τονίσω, ακριβώς αφορά αυτό που ήθελα να αναφέρω, είναι οι κανόνες του ΠΟΕ, όπου μέχρι στιγμής δημιουργούν πλήρες αδιέξοδο και στην πτυχή των κλιματικών αλλαγών. Βλέπουμε δηλαδή ότι χρειάζεται να ληφθούν, ναι, να ληφθούν αποφάσεις πάνω σε αυτό το τομέα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού για το περιβάλλον. Πέμπτο μου σημείο και καταλήγω μετά στο ποια θα πρέπει κατά την άποψή μου να είναι η δική μας οπτική για το εμπόριο. Πέμπτο σημείο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενσωματώσει σε όλες τις εμπορικές συνδιαλλαγές και στις εμπορικές συμφωνίες και μια ρήτρα για το περιβάλλον. Μια ρήτρα που σχετίζεται με την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος και μας δίνεται η ευκαιρία εφόσον με τη μεταρρύθμιση του καταστατικού ΖΕΣΠΕΣΙΝ θα έχουμε τη δυνατότητα εδώ στην Επιτροπή Ανάπτυξης να επιβάλλουμε την ενσωμάτωση ενός κλιματικού κριτηρίου σε αυτό το καταστατικό. Σας ευχαριστώ και είμαι διαθέσιμη να ακούσω τις παρατηρήσεις σας πριν να σας παρουσιάσω λίγο αργότερο τροποποιήσεις ε, προς την κατεύθυνση που σας ανέφερα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχουν οι βουλευτές. Τώρα, ο κύριος Αρσένης πρώτα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, Βρίσκω την γνωμοδότηση πολύ καλή, ε, πραγματικά κινείται στη σωστή κατεύθυνση και συμφωνώ μαζί τους. Το μόνο που ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι θα ήθελα να γίνεται πιο συγκεκριμένη ε, αναφορά στην προσαρμογή σε σχέση με την ε, ε, των, των διατάξεων. Ίσως να υποβάλω κάποια τροπολογία σε σχέση με αυτό. Εν γέννη πάντως η έκθεση είναι πολύ καλή και κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Επιτροπή, την οποία εκπροσωπεί ο κύριος Ούλρικ Βάιγκελ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Παύλος Καλίδης είμαι από την Επιτροπή. Ε, ο κύριος Βάγκελ δεν μπόρεσε να είναι εδώ και θα μιλήσω στα αγγλικά. Το πρώτο που θέλω να πω αφορά τα σημεία που αφορούν τις επιπτώσεις του εμπορίου στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Φυσικά δεν υπάρχει αμφιβολία περί αυτού ότι υπάρχει δηλαδή άμεση σχέση, ωστόσο θα πρέπει να εξετάσουμε και άλλε πτυχέ ιδιαίτερα το θέμα της σύσταση, δηλαδή ότι η παραγωγή κινείται προ πιο επαρκεί παραγωγού. όσον αφορά την εκπομπή δηλαδή αερίων του θερμοκηπίου, γιατί αυτό προωθείται και από το εμπόριο και από τον ε, ε, ανταγωνισμό. Ε, καλύτερη πρόσβαση επίσης στις κλιματικές τεχνολογίες υπάρχει ήδη. Γενικά νομίζω πως χρειάζεται να υπάρχει μια γενική ανάλυση, τα, ας πούμε ότι η τοπική παραγωγή και κατανάλωση είναι πάντοτε η καλύτερη σε θέματα εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου και διοξιδίου του άνθρακα, αλλά δεν είναι πάντοτε αυτονόητο και πρέπει αυτό να εξεταστεί. Παρόμοια παρατήρηση σε σχέση με τη γεωργία και πάλι ναι, υπάρχει βέβαια βάση στα όσα λέγονται, αλλά και πάλι χρειάζεται ανάλυση του πλήρους κύκλου ζωής για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε έγκυρα αποτελέσματα όσον αφορά το κόστος ε, παραγωγής σε διάφορα μέρη του κόσμου. Εξίσου θα πρέπει να εκτιμήσουμε κατά πόσο η προώθηση της οργανικής καλλιέργειας μήπως δημιουργήσει προβλήματα ασφάλειας στα τρόφιμα για ορισμένες χώρες. Παράγραφος 3. Αγορές. Εδώ έχουμε διαφορετική εκτίμηση για το κατά πόσο δουλεύουμε, για το πώς μάλλον θα πρέπει να δουλέψουμε ή όχι. Αν, όσον αφορά το ευρωπαϊκό σύστημα πορεία εκπομπών πιστεύουμε ότι δουλεύει, ότι λειτουργεί και ότι δεν υπάρχει λόγος να ε, γίνει παρέμβαση στις τιμές ή στο να περιοριστούν οι τιμές. Εγώ ήθελα να ξέρω ποιες ακριβώς είναι οι ανησυχίες του εισηγήτριας για αυτό το θέμα. Μιλήσατε για το θέμα της ε, πτυτικότητας των τιμών, της, μετα... της ε, ε, και αυτό υπάρχει και λειτουργεί ότι, σημαίνει ότι λειτουργεί σωστά η αγορά κάθε φορά. δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο στόχος μας είναι να έχουμε ε, μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και με καλό κόστος. Και γενικά λοιπόν πιστεύουμε ότι το σύστημα λειτουργεί καλά. Τώρα, για την διαρροή άνθρακα δεν χρειάζεται να μιλήσω πολύ γι' αυτό, γιατί η Κομισιόν έχει κάνει μια ανακοίνωση θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι, ποιες θα είναι οι δυνατότητες ε, που μπορούμε να επιτρέψουμε για την επόμενη περίοδο 2020-2030. Θεωρούμε πως ε, κλειδί για τη λύση αυτού του θέματος είναι μια διεθνή συμφωνία για το κλίμα. Ε, δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ελπίζουμε ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Και βεβαίω θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε τα συνοριακά μέτρα ως επιλογή για το μέλλον, αλλά αυτή είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή που θα εξετάσουμε. Θα μπορούσα να κάνω και μια παρατήρηση για τον ε, ΠΟΕ και για τις διμερείς συμφωνίες, για το GPS-SYN, ε, το Kyoto, η και το πρωτόκολλό του, μάλλον και η συνεπογραφή του πρωτόκολλου του είναι προϋπόθεση και σίγουρα εμείς θέλουμε να θέσουμε νέους όρους που σχετίζονται με το περιβάλλον σε ένα, στο νέο καθεστώς GPS. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Γκρέσ έχετε εκ νέου το λόγο. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Άκουσα με προσοχή τις παρατηρήσεις που έγιναν ιδίω όσον αφορά την αναγκαιότητα να ληφθούν υπόψη ε, την ανάγκη λέω να ανεπτυχθεί το θέμα και όσον αφορά τη γεωργία και τις σχέσεις μεταξύ της ε, ε, ασφάλειας αφενός και της ε, βιολογικής γεωργίας αφετέρου. Προς τον συνάδελφο της Κομισιόν Έχω να πω ότι τα σχόλια του δίνουν εντύπωση ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει μία ρήτρα για το περιβάλλον. Χρειάζεται όμως. Χρειάζεται να έχουμε αυτό που το αποκαλούμε capacity building. Νομίζω όμως και το τονίζεται αναφερόμενο στο πρωτόκολλο του Κιώτο που έχει στο στόχο να δυναμωθούν οι περιβαλλοντικές πτυχές Πιστεύω, λέω, ότι αν θέλουμε πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση στις εμπορικές σχέσεις να λαμβάνει υπόψη τα θέματα των κλιματολογικών αλλαγών και των, της περιβαλλοντικής ψυχές, θα πρέπει να παραβλέψουμε την ανάγκη μια τέτοια ρήτρα. Αυτό νομίζω είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο σημείο 8 τη ημερησία διάταξη. Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτο που εφαρμόζει το λοιπό προσωπικό των κοινοτήτων. Έγκριση απόφαση του Συμβουλίου όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία ε, των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απόφαση που λήφθη ε, Υπουργού 26 Ιουλίου 2006 και για την οποία υπάρχει μια σκέψη της 9ης Ιουλίου του περασμένου έτους και που θα εξαστεί αυτή την εβδομάδα στην Μαδρίτη. Για να μπορεί η εξωτερική υπηρεσία να είναι λειτουργική χρειάζονται ακόμα προσαρμογές στον ε, ε, δημοσιονομική πτυχή και το καθεστώς του των υπαλλήλων. Αυτές είναι οι δύο πτυχές που μας ενδιαφέρουν. Πρόκειται για δύο νομιθικά σφακέρους που εξετάζονται αυτή τη στιγμή. Σήμερα θα ψηφίσουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για πάνω στην έκθεση της Επιτροπής των Προεπολογισμών όσον αφορά την τροποποίηση του ε, δημοσιονομικού κανονισμού. Τώρα θα εξετάσουμε την πρόταση ψηφίσματο του συνάδελφου Φίλιπ Κασμαρέκ πάνω στην έκθεση του κυρίου Μπέρνατ Καράπκη για την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Φίλιπ Κασμαρέκ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να πω ότι η έκθεση του κυρίου Ραπκάη κατά τη γνώμη μας είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς εδώ στην Επιτροπή μας μπορούμε απόλυτα να υποστηρίξουμε την έκθεση χωρίς να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Τρία θέματα θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με την ε, έκθεση Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Καταρχήν, θα πρέπει να συμφωνήσουμε Ε, η απόσπαση του προσωπικού για την υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων να γίνει με διαφανή τρόπο. Αυτό νομίζω είναι κάτι που μπορούμε να βρούμε σύμφωνος. Επίσης θα πρέπει να συμφωνήσουμε νομίζω να έχουμε μια πιο σύντομη ε, προθεσμία από την οποία και μετά το προσωπικό του κοινοβουλίου μπορεί να ζητήσει να ενταχθεί <clears throat> στην υπηρεσία αυτή. Η Κομισιόν λέει 1η Ιουλίου 2013. Ο κ. Ζαπκάια αναφέρεται στην 1η Ιανουαρίου 2012. Ένα μισό χρόνο πριν δηλαδή. Δηλαδή θα μπορέσουν να ανοίξει αυτή η ιανουαριου 2012 ενα μισο χρονο πριν δηλαδη δηλαδη θα μπορεσει να ανοιξει αυτη η διαβλωση για το προσωπικό της Κομισιόν και του ε, Κοινοβουλίου ένα μισό χρόνο πριν από ό,τι προτείνει η ίδια η Κομισιόν. Επίσης θα πρέπει να έχουμε μια αναφορά στην ε, ισορροπία ε, φύλων αλλά και τη γεωγραφική ισορροπία. Η διατύπωση είναι πάρα πολύ σαφής. Αυτό που λέω εγώ οπωσδήποτε ήταν καινούριο. Είναι θέματα που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Όταν συζητάγαμε την εγκαθίδρυση της υπηρεσίας για τις εξωτερικές δράσεις, ε, η πρόταση μου περιλαμβάνει δύο τροπολογίες. Η πρώτη αφορά τον ορισμό των διπλωματικών υπηρεσιών, γιατί αναφερόμαστε στις ε, διπλωματικές υπηρεσίες των κρατών μελών. Χρειαζόμαστε όμως πιο ευρύ ορισμό, ούτω ώστε να καλύψουμε όλο το προσωπικό που ασχολείται στις υπηρεσίες αυτής ασφάλεια, άμυνα, ανάπτυξη προστασία του περιβάλλοντος και εξωτερικό εμπόριο. Δηλαδή, αυτό που εννοώ είναι ότι το διπλωματικό προσωπικό που ασχολείται με την ανάπτυξη θα πρέπει να μπορεί να ζητήσει να ενταχθεί στην υπηρεσία εξωτερικών δράσεων της Ένωσης. Η δεύτερη μου τροπολογία αφορά την ενδυνάμωση του ρόλου του αρμοδίου εκάστοτε επιτρόπου. όσον αφορά τα ανθρωπιστικά θέματα. Είναι κάτι που νομίζω το συζητήσαμε ήδη όταν εξετάσαμε το θέμα της ε, εγκαθίδρυσης της υπηρεσίας αυτής δράσεων. Νομίζω θα παίξει ο ρόλος της ε, ε, Κομισιόν να είναι πιο έντονος, δεν φαντάζομαι να διαφωνήσει κανένας με αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Τώρα σας ευχαριστώ. βουλευτές έχουν το λόγο τώρα. Ο κ. Γκερέρο θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ραπκάη, συγκεκριτή εξουσία για την έκθεσή του και θα ήθελα επίσης να συμφωνώσω με κάποιες από τις συστάσεις που παρουσίασε ο κύριος Κάσπαρέκ. Είναι πραγματικά πολύ καλό θα επιμείνουμε το καθεστώς των υπαλλήλων να συμπεριλαμβάνει, να καλύπτει μάλλον τους περισσότερους κατά τα που αναλαμβάνουν κάποιο έργο εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανά τον κόσμο. Είναι σημαντικό και το είπανε διάφοροι από εμά στο παρελθόν σε μια συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναπτυξιακή Βοήθεια ότι είναι λέω σημαντικό να υποστηρίξουμε και το ρόλο του αρμοδίου επιτρόπου. Να τονίσουμε το θέμα της ορατότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ. La parole est au cabinet de Madame. Το λόγο έχει εκπρόσωπο του εσωτερικού γραφείου της κυρίας Άστον, στον κύριο Παουλ Κριστόφερσον. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας αποτείνω το λόγο στην Επιτροπή σας. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για το σωματικό έργο που επιτελέστε στην προετοιμασία της γνωμοτότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον βασικό κανονισμό που υιοθετήθηκε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία τον Ιούλιο θα είδατε φαντάζομαι ότι πολλές από τις τροπολογίες που πρότεινε η Επιτροπή Ανάπτυξης εντάχθηκαν τελικά στη βασική απόφαση. Επίσης είναι σαφές ότι παρόλο που αυτή η αρχική απόφαση ήταν ότι χρειάζεται μόνο μια αγνομοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τελικά de facto καταλήξαμε σε συναπόφαση. Και η γνωμοδότηση που ευθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούλιο αντικατοπτρίζεται λέξη προς λέξη στην τελική απόφαση του Συμβουλίου του Ιουλίου. Βάσει αυτών είναι πάρα πολύ σημαντικό Αυτό που γίνεται όσον αφορά τις απαραίτητες αλλαγές στον δημοσιονομικό κανονισμό και στον κανονισμό ε, υπηρεσία κατάστασης των υπαλλήλων αντικατοπτρίζουν απόλυτα, λέω, τα αποτελέσματα των Ιουλίου. Δεν θέλω να αναφερθώ στο ερώτημα που έθεξε ο κ. Κασμαρέκ. Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με την έντυπωσή του ότι δηλαδή η έκθεση του κ. Ραπκάη αποτελεί πάρα πολύ καλή βάση για συμφωνία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Ελπίζουμε στην πρώτη ανάγνωση ήδη. Και σύντομα. Α, όσον αναφέρεται το θέμα της διαφανούς πρόσληψης κλπ. Οπωσδήποτε συμφωνούμε απόλυτα. Και αυτά είναι θέματα που έχουμε ήδη συζητήσει στο παρελθόν. Υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ημερομηνία για προσλήψη από τα άλλα θεσμικά όργανα, γιατί η συμφωνία του Ιουλίου όριζε μια συγκεκριμένη ημερομηνία που ήταν 2013, τέλη 2013. Είναι δύσκολο τώρα να το αλλάξουμε αυτό. Όσον αφορά τα δύο συγκεκριμένα θέματα που εθίγησαν στο σχέδιο της γνωμοδότησης, έχω να πω τα εξή. Στο πρώτο, όσον αφορά το θέμα του ορισμού του διπλωματικού σώματος. Θα μπορούσα να συμφωνούσα βάσει αυτό που είπε ο κ. ότι θα πρέπει να έχουμε κατά τον ευρύ ορισμό τι είναι η διπλωματική υπηρεσία. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν όρια. Τα όρια είναι η συνθήκη, η οποία είναι αρκετά ακριβής για το θέμα αυτό. Και φοβούμαι ότι αν τελικά είχαμε τόσο ευρύ ορισμό όσο αναφέρεται στο άρθρο 1, υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθούμε σε αντίφαση με την ίδια τη συνθήκη. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί βέβαια αυτό είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε στο μίσο που ξεκινήσαμε τη διαδικασία πρόσληψης δίνοντας de facto στις ε, εθνικές αρχές <clears throat> ε, ευρύ, φάσμα να αποφασίσουν μέσα σε αυτό τι θεωρούν οι ίδιοι διπλωματικό σώμα. Το δεύτερο τώρα, όσον αφορά το προγραμματισμό, ότι γίνεται από την ΙΕΣ δηλαδή, και κατόπιν μια πρόταση από την Επιτροπή Ανάπτυξης. ότι θα πρέπει να είναι αυτό υπό την ευθύνη του Επιτρόπου που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη. Αυτό νομίζω είναι κάτι που θα γίνει στο ΙΕΣ. E Γιατί ε, το 1,9 που έχουμε εδώ αναφέρει το τι έχει γίνει στις διάφορες αντιπροσωπείες και τι γίνεται όσον αφορά το τελευταίο στάδιο το οποίο είναι υπό την ευθύνη της Κομισιόν. Γι' αυτό λοιπόν δεν είμαι καθόλου σίγουρος κατά πόσο αυτή η προστίκη χρειάζεται στο κείμενο. Αυτά είχα να πω πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον κύριο Κεσολάκη, αν το διάβασα καλά το όνομά σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μπορώ να συμφωνήσω με τον εκπρόσωπο τη ΥΠΑ του εκπροσώπου και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά που είπε. Θεωρούμε πράγματι ότι θέματα ισορροπία μεταξύ των φύλων και γεωγραφική ισορροπία είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και υπάρχει ευρεία συμφωνία πάνω σε αυτά που προτείνει ο κ. Ραπκάη. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, θα θέλαμε να πούμε ότι αυτό θα πρέπει να λειτουργεί και ε, στις δύο ομάδες, δηλαδή και στους ε, και στους υπευθύνους και στο βοηθητικό προσωπικό. Επίσης συμφωνούμε ότι ο... να αλλάξει η ημερομηνία αντί 1η Ιουλίου 2013 να λέμε 1η 2012 τότε θα είναι πολύ δύσκολο η υπηρεσία εξωτερικής δράσης να ε, εξασφαλίσει σωστή εκπροσώπηση ε, εθνικών διπλωματών, τα κρατημέλη δηλαδή, που είναι ένας όρος. Η Κομισιό πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει μόνο σε τρία χρόνια πριν από την πρώτη εβδόμου, δηλαδή 2013. Και όσον αφορά τις που προτείνει η Επιτροπή σας, το ορισμό του πνευματικού σώματος. Αυτό δεν είναι θέμα του κανονισμού υπηρεσιακής ε, κατάστασης. Αυτός ο κανονισμός ασχολείται με τις σχέσεις μεταξύ του προσωπικού και των θεσμικών οργάνων. Και εγώ πιστεύω ότι τα υπόλοιπα θα πρέπει να οριστούν από την απόφαση του Συμβουλίου που εγκαθιδρεί την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Όσον αφορά τη δεύτερη προτενόμενη τροπολογία, Πιστεύουμε ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και να παραβλέπουμε την απόφαση που εγκαθιδρεί την Υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα πρέπει να την... αυτό που λέτε εδώ όμως να μην το έχουμε στο κείμενο μάλλον να το έχουμε μάλλον στις ιδεολογικές σκέψεις. Γιατί ένας υπάλληλος Επιτροπής Εξωτερικών ε, ε, Δράσεων θα πρέπει να δράσει βέβαια βάσει κάποιων κατευθυνών γραμμών της Κομισιόν χωρίς να αναφέρει τις κατευθυντήρες αυτές ρητά. Αυτό αναφέρει σε άλλο κείμενο. Ευχαριστώ αυτά. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαρεκ. Αν θέλετε, έχετε το λόγο να ολοκληρώσετε. Ναι, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, είμαι ευγνώμων για τα διάφορα σχόλια που άκουσα. Η ιδέα όσον αφορά διατύπωση σχετικά με το διπλωματικό σώμα είναι να είμαστε σίγουροι ότι το προσωπικό των πολιτικών ανάπτυξης μπορεί να δραστηριοποιηθεί μέσα στα πλαίσια της υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Ίσως ε, αυτό που λέμε η διατύπωση και άλλες πολιτικές ίσως είναι πολύ ευρεία, αλλά εγώ θεωρώ ότι το προσωπικό που ασχολείται με την ανάπτυξη θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί γιατί η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων καλύπτει ακριβώς αυτό το Για τη δεύτερη τροπολογία. Και εδώ η πρόθεση είναι να εξασφαλίσουμε ο Επίτροπος να έχει κάποια επίδραση πάνω στο πώς λειτουργεί η υπηρεσία εξωτερικών δράσεων. Να εξασφαλιστεί δηλαδή η συνεργασία μεταξύ των προσωπιών και της Κομισιόν, γιατί θα πρέπει να συνεργαστούν. μα όσον αφορά τη χρηματοδότηση, τον προγραμματισμό κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι υπό την ηγεσία τη Κομισιόν. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ. Σα ενημερώνω ότι η προθεσμένη νομοβολή των απολογιών είναι Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου στι 12 το μεσημέρι και η ψηφοφορία στην Αρμόδια Επιτροπή θα γίνει στην επόμενη μα τακτική συνεδρία στι 4 και 5 Οκτωβρίου. Περνάμε τώρα στην τροποποίηση του κανονισμού 1905-2006 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση επιγονισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας. Λίγο πριν από τι κοινοβουλευτικέ διακοπέ, είχαμε μια πρώτη ανεπίσημη συζήτηση πάνω στην πρόταση τη Κομισιόν για μια τροποποίηση του μέσου χρηματοδότηση τη συνεργασία για την ανάπτυξη, του DCI, για να μπορέσει να προσθεθεί ένα νέο πρόγραμμα που αφορά μέτρα συνοδευτικά για τον τομέα της μπανάνας υπέρ των κυρίων χωρών και παραγωγής μπανάνας βάσει των, της μείωσης των ε, δεδομενικών προτιμήσεων που δόθηκε στις χώρες αυτές. Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν μία ενίσχυση 190 εκατομμυρίων συγγνώμη, ευρώ σε 4 χρόνια σε 10 χώρες παραγωγούν πανάνας ιδίως αυτών που έχουν πληγεί από την συμφωνία που επιτέχθηκε μέσα στα πρέσια του ΠΟΕ. Η Επιτροπή μας είναι αρμόδια της ουσίας για την νομοθετική έκθεση πάνω στην πρώτη αυτή. Και ο εισητής μας είναι ο κύριος ε, Γκόρενς. Θα δείτε ότι ο κύριος Γκόρενς δεν ήταν αργός προς κατά των διακοπών, θα του δώσω αμέσω το λόγο να σα παρουσιάσει την έκθεση που προετοίμασε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, τα πράγματα έχουν ε, κάπως ε, περιπλακεί, αλλά η ουσία μένει. Αυτό το οποίο εμάς ε, μας ανησυχούσε εδώ στην Επιτροπή ήταν να μπορέσουμε να μείνουμε ε, συνεπής ε, στην καταπολέμηση της στόχιας ε, και από αυτή την οπτική εγώ με την στήριξή σας ε, υποστηρίζω αυτά τα μέτρα που στόχο έχουν να αντισταθμίσουν τις επιπτώσεις μιας εμπορικής συμφωνίας ε, που είναι τέτοιας φύσης ώστε να επιδεινώνει κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση των ε, εξαγωγών των εξαγωγών μπανάνας των χωρών της Αφρικής και του Ειρηνικού. Πρόκειται για καμιά δεκαριά χώρες. και υπ' αυτές τις επιφυλάξεις ε, σας ε, υποβάλλω τις τροπολογίες που έχετε. Καταρχήν, ε, κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά τον γύρο της Ντόχα για την ανάπτυξη που είχε τη φιλοδοξία να λάβει υπόψη την ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Σε δεύτερον, Κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε από τη μελέτη που είχαμε εκπονήσει εδώ στην Επιτροπή μας και που αφορούσε την διαδρομή της μπανάνας που μας οδήγησε στο να καταλήξουμε ότι ο παραγωγός είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τα λιγότερα από ολόκληρο το ποσό που συγκεντρώνεται κατά τη διάρκεια της πορείας που διανύει η μπανάνα από τον αρχικό της παραγωγό μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οι άλλες τροπολογίες θα πρέπει να εξεταστούν υπό την ίδια οπτική γωνία. Φυσικά περιμένω με ανυπομονησία τις αντιδράσεις των μελών της Επιτροπής μας και επίσης τις αντιδράσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία αυτού του εγγράφου. Η τροπολογία που αποτελεί την καρδιά της έκθεσής μας είναι η τροπολογία που αφορά το άρθρο 17. Αφορά τη στρατηγική πολιετούς ε, αρρωγής για την στήριξη της μπανάνας. Σε προηγούμενες συνεδριάσεις επιμείναμε ότι ο βασικός μας στόχος είναι η καταπολέμηση της στόχιας. Αυτή η καταπολέμηση της στόχιας θα πρέπει να βασίζεται στην ε, πραγματικότητα επιτόπου. Δηλαδή θα πρέπει να θέτουμε στόχους οι οποίοι να είναι μετρήσιμοι, μετρήσιμοι στο μέτρο του θυνατού και οι οποίοι θα πρέπει να υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να δούμε πως η αξιολόγηση θα πρέπει να αποτελεί στο τμήμα ενός αναπτυξιακού προγράμματος και θα πρέπει μάλιστα να κατέχει τιμητική θέση στην αρχή ενός κύκλου προγραμμάτων. Θα πρέπει δηλαδή οι όροι αναφοράς για την αξιολόγηση να είναι γνωστή από την αρχή ενός κύκλου προγραμματικού. Και από αυτή την οπτική γωνία θα πρέπει να αναλύσουμε την τροπολογία αυτή, όπου καλούμε κυρίως και νομίζω πως αυτή ήταν μια παρατήρηση που έκανε η κυρία Κρές τις επιπτώσεις των ζυζανιοκτώνων στα φρούτα αλλά και στους ανθρώπους, στους καρπούς αλλά και στους ανθρώπους που εργάζονται ε, σε αυτό το τομέα. Ε, περιβαλλοντικό προφίλ της χώρας ε, και μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος στον τομέα της παραγωγής μπανάνας. Αν θέλουμε να είμαστε λοιπόν συνεπείς στο στόχο μας θα πρέπει να συμπεριλάβουμε το στοιχείο αυτό που έχει την ε, περιβαλλοντική διάσταση και που αφορά και την υγεία των παραγωγών. Β. Αυτό που είπα μόλις, ότι δηλαδή ζητάμε προδιαγραφές για την ε, ανεξάρτητη αξιολόγηση των μέτρων εφαρμογής. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τι ακριβώς θα αξιολογηθεί, με βάση αυτή τη συμφωνία, καθώς και όρους επιλεξιμότητας σε περίπτωση δημοσιονομικής στήριξης, για τη δυνατότητα δηλαδή παροχής ε, ενίσχυσης. Το τρίτο σημείο αναφέρεται σε μια συζήτηση για τη μορφή που μπορεί να έχουν οι διάφορες ενισχύσεις. Υπάρχουν χώρε οι οποίες θα ωφεληθούν από αυτά τα μέτρα και που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προϋπολογισμού τους, μέσω του δημοσιονομική της δημοσιονομικής στήριξης και εκεί θα ήθελα να γνωρίζω ποιε είναι οι απόφασεις. Ακόμα και αν δεν εξαρτάται από την χώρα δέκτη, τη χώρα δικαιούχου, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα χρήματα τα οποία προορίζονται για την αντιστάθμιση ενός μειονεκτήματος που προκύπτει από μία εμπορική συμφωνία θα φτάνουν ακριβώς στους ανθρώπους οι οποίοι πλήττονται από τη συμφωνία. Δηλαδή, ακόμα και αν τα χρήματα κυκλοφορούν μέσα από τον προϋπολογισμό της χώρας που τα λαμβάνει, θα πρέπει ο αντίκτυπος των χρημάτων αυτών να ε, μπορεί να μετρηθεί. Γιατί εάν δεν υπάρχει τέτοια κατάληξη δεν κάνουμε σωστή δουλειά. Τέλος, ε, τα αποτελέσματα που περιμένουμε για το τομέα της μπανάνας μετά από συγκεκριμένες δράσεις θα είναι σημαντικό να παρακολουθηθούν. Ο τομέας της μπανάνας θα περάσει από μεγάλες ε, μετατροπές. Στόχος είναι να είναι πιο αποδοτικός ο τομέας. Αν κάτι τέτοιο δεν είναι δεδομένο θα πρέπει να γίνει αναδόμηση, αναδιάρθρωση να δούμε, εν πάση τι μπορούμε να κάνουμε με μέσα τα οποία ε, θα πρέπει να οδηγήσουν στην ε, μετατροπή, στην αναδιάρθρωση. Αυτά αποτελούν τμήμα της λογικής την οποία υιοθετήσαμε στις προηγούμενες μας συνεδριάσεις. Έπειτα, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις μεταρρυθμίσεις και για τις δαπάνες για κάθε δικαιούχο χώρα. Καθώς η Κομισιόν θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί με κάθε χώρα δικαιούχο ενίσχυσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα των μεταρρυθμίσεων και βεβαίως <coughs> τις προβλέψεις για τις δαπάνες για κάθε δικαιούχο χώρα. Το F αφορά τον κατάλογο και τις προδιαγραφές του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ώστε να προστατευτεί η υγεία των εργαζομένων. Η στρατηγική αυτή αποτελεί αντικείμενο μιας ανεξάρτητης ε, αξιολόγησης και σε περίπτωση που αυτό χρειάζεται μιας επιτόπου, ενός επιτόπου ελέγχου. Και εδώ, ο Διεθνή Οργανισμό Εργασία, αν θέλει να έχει νόημα ύπαρξη, θα πρέπει να σταθεί στο πλευρό των πιο φτωχών και των πιο ευάλωτων. Και με αυτή την έννοια εισάγαμε αυτήν την τροπολογία, ώστε οι προσανατολισμοί και οι κανόνες που ορίζει ο, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας να μην μείνουν νεκρό γράμμα. Αυτά κατά βάση. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα συζητάμε, γι' αυτό και δεν θα σας αναφέρω όλες τις πτυχές ε, ε, που έχουν αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων μας συζητήσεων. Να προσθέσω επίσης, και εδώ νομίζω μπορούμε να ωφεληθούμε από αυτήν την έκθεση και να την εκμεταλλευτούμε, ώστε να πούμε ότι στο πλαίσιο των ε, πόρων που πηγαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες έχουμε πρόβλημα. Έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο μας τόνισαν οι ΜΚΟ. Ότι δηλαδή οι φόροι και κυρίως ο ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που πρέπει να καταβληθεί για ένα αντικείμενο το οποίο πάει στην, ε, στις χώρες αυτές δικαιούχους βοήθειας δεν μπορεί να αποτελέσει, να επιβαρύνει μάλλον ε, τον κοινοτικό προπολογισμό. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να τελειώσει πια αυτή η αδικία. Για τις ΜΚΟ οι οποίες εκπληρούν ε, μεγάλη αποστολή γιατί πρέπει περισσότερο να ασχοληθούν με τη συλλογή κονδυλίων και όχι με την δουλειά για την οποία βρίσκονται εκεί. Και αυτό μου φαίνεται πως είναι αδύνατο. Είναι ένας φόρος ο οποίος είναι μια δαπάνη, αν και σε επίπεδο της κοινοτική ορθοδοξίας δεν έχει ε, δημιουργεί μόνο ένα ε, πρόβλημα, ένα πρόσκομα. Θέλω να καλέσω λοιπόν την Επιτροπή να το σκεφτεί αυτό πολύ πολύ σοβαρά. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Οι ευρωβουλευτέ τώρα έχουν το λόγο. Κυρία Κρέση, έχετε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε στις διακοπές και για την έκθεση που μας παρουσίασε. Τον ευχαριστώ επίσης πολύ που εισακούστηκαν οι προτάσεις των πρασίνων για την προστασία του περιβάλλοντος και κυρίως όσον αφορά την υγεία των ανθρώπων που δουλεύουν στην μπανάνα, που εκτίθενται μαζικά στα παρασιτοκτόνα. Πάντως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε κάποια σημεία παρόλα αυτά. Για το θέμα της εντατικής καλλιέργειας μπανάνας, χωρίς αλλαγή, γιατί Πάντα υπάρχουν θέματα που παραμένουν σε κρεμότητα, όπως είναι το ότι το έδαφος χάνει τις πλούσιες ουσίες του. Και κάτι ακόμα που θέλω εδώ να αναφέρω είναι περισσότερο προς ε, τα μέλη της Επιτροπής μας. Δεν είμαι σίγουρη, το λέω από την αρχή. Άκουσα ότι οι Υπουργοί Καμερούν, Γκάνα και Ακτήλε Φαντοστού συζήτησαν μεταξύ τους για να συζητήσουν το πρόγραμμα και μας έκαναν την εξής παρατήρηση ότι πρόκειται για το τελευταίο σχέδιο που είναι υπέρ της μπανάνας, μας είπαν. Αλλά αυτή είναι ερώτηση από τη δικιά μου την πλευρά. Είναι έτσι ή όχι. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι έχουν ληφθεί υπόψη οι παράγοντες υγεία και περιβάλλον στο κείμενο αυτό. Πρέπει πάντα να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι μοντέλο καλλιέργειας χρησιμοποιούμε για την παραγωγή μπανάνας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Πόγκα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Γκέρενς για την εξαίρετη δουλειά του. Είναι ένα πολύπλοκο θέμα. Τι διακυδεύεται όσον αφορά την ανάπτυξη των χωρών ΑΚΕ που παράγουν μπανάνα. Είναι τεράστια αυτά που δακυδεύονται. Πρώτα απ' όλα είμαστε οι πρώτοι και παραγωγοί και καταναλωτές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ιδιαίτερε σχέσει, προνομιούχε με τι χώρε ΑΚΕ. Όσον αφορά τώρα το σχέδιο κειμένου του κ. Γκέρεν, πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ότι παραμένουν κάποια σημεία. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική που προτείνουμε πιο μακροπρόθεσμη και όχι βραχυπρόθεσμη, χωρίς να υπάρχει η προοπτική για η φόρο ανάπτυξη. Η Επιτροπή στο σχέδιο κανονισμού της προβλέπει μέτρα προσωρινού χαρακτήρα, τεσσάρων ετών κατανότατο, μέχρι το 2013 δηλαδή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις συνέπειες των διμερών συμφωνιών που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και που προβλέπουν δασμολογική μείωση πιο μεγάλη από αυτήν που προβλέπεται στη Συμφωνία της Γενέβης. Ορισμένε χώρε χώρες της Λατινικής Αμερικής, για παράδειγμα, που είναι κύριοι παραγωγή μπανάνα παγκοσμίω. Επίση, πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ λιγάκι και τα κριτήρια για τη χορήγηση βοήθεια. Η βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βασίζεται σε σαφή κριτήρια και σωστά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση αυτή να διέπεται από διαφάνεια. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια στάθμιση στους δείκτες τους οποίου χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καθορίσει το ποσό των ενισχύσεων. Αυτή η στάθμιση υπογραμμίστηκε και στη διάσκεψη της Γιαουντέ στις 23 Ιουλίου που μας πέρασε, όπου συναντήθηκαν οι Υπουργοί Εμπορίου του Καμερούν, της Ακτής Ελεφαντοστού και της Γκάνα. Οι κύριες αφρικανικές χώρες που παράγουν μπανάνα, όπως πολύ σωστά είπαμε. Τέλος, πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση και συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο των χωρών και αυτό πρέπει να το πούμε όταν μιλάμε για την παραγωγή μπανάνας και κυρίως σε σχέση με τις άκρος περιφερειακές περιοχές. Δεν πρόκειται για την Καραϊβική ή Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Στυρολίαν θέλει το λόγο τώρα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον εισηγητή μας για την δουλειά του. Έτσι σήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ένα κείμενο ποιότητας. Όμως θέλω να επανέλθω σε μερικά σημεία που πιστεύω ότι είναι σημαντικά και πιστεύω ότι μπορούν να βελτιώσουν το κείμενο. Το πρώτο μου σημείο έχει να κάνει με τον τρόπο χρηματοδότησης του μέσου αυτού. Έχουμε μαθήματα από προηγούμενους κανονισμούς του 94, του 99. Εμπειρία πολύτιμη για να μας βοηθήσει στο μέλλον. Τόσο στην περίπτωση 1994 που μιλούσαμε για τα έσοδα και του 99 που έδινε πρόσβαση σε προγράμματα επενδύσεων και τα δύο κατέληξαν σε καταστροφή μειώθηκε η ανταγωνιστικότητα των χωρών παραγωγών ε, ΑΚΕ εξαιτία του ΠΟΕ. Η καλή στρατηγική λοιπόν είναι να δεχτούμε την ευελιξία και να στηρίξουμε τους παραγωγούς ανάλογα με τη συμπεριφορά της αγοράς. Δεν είναι αυτό όμως που έχει επιλέξει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την πρότασή της. Το δεύτερο σημείο που πιστεύω ότι είναι επίσης σημαντικό και ο κύριος Πόγκα λίγο πολύ αναφέρθηκε σε αυτό, είναι η κατανομή των ε, πόρων στις διάφορες χώρες, ξεκινώντας από κάτω. Η κατανομή αυτή δεν διέπεται από διαφάνεια. Υπάρχουν τρία κριτήρια που έχουν επιλεχθεί από την Επιτροπή, αλλά η Επιτροπή δεν μας μιλάει καθόλου για τον συντελεστή που θα μας επιτρέψει να έχουμε σωστή αξιολόγηση ενώ οι αφρικανικές χώρες ολοκληρώνουν το δικό του σχέδιο που είχε προθεσμία 10 έτη, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία πρόβλεψη βάσει της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έτσι δεν μπορούν οι χώρες αυτές να ετοιμάσουν μια νέα στρατηγική που να αξίζει το όνομά της. Αυτά είχα να σας πω και βάσει αυτών θα φροντίσω να υποβάλω και τροπολογίες στον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τώρα το λόγο. Ο κύριος Βίμ Χολτχοφ εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ πολύ που μας επιτρέπετε να μιλήσουμε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Ευχαριστούμε τον κύριο Κέρενς και τους συνεργάτες του για την υψηλή ποιότητα του κειμένου που ετοίμασε. Πρέπει εδώ να σας πω ότι στην εσωτερική διαδικασία διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που βέβαια καταλαβαίνετε διακόπηκε με τις καλοκαιρινές διακοπές, είμαστε ακόμα στην αρχή. Εγώ θα αναφερθώ σε 8 σημεία. Πρώτα απ' όλα, χαίρομαι πολύ που στην έκθεση αυτή και που στην αιτιολογική σκέψη αναφέρονται όλες οι βασικές πτυχές που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις υποστηρίζει από ό,τι βλέπω ο εισηγητής σας. Οπότε είναι καλό αυτό. Δεύτερον όμως, σημειώνουμε ότι το σχέδιο έκθεσης περιλαμβάνει 14 τροπολογίες, 5 από τις οποίες προτείνουν να μιλήσουμε για τις κατεξουσιοδότηση πράκτηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη υποβάλει αντίστοιχες ε, τροπολογίες και στα πλαίσια της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης για την εξωτερική χρηματοδότηση. Οπότε ανεξάρτητα από το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συμμερίζεται τι απόψει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να θεωρηθούν κατά εξουδότηση πράξει στρατηγικέ αυτέ, παρόλα αυτά οι τροπολογίε δεν χρειάζεται να βρίσκονται εδώ. Επιπλέον, η συζήτηση για την φύση των προγραμμάτων σε κείμενα στρατηγική και όσον αφορά το κατά πόσο εφαρμόζεται τα 290 και 291 τη συνθήκη που αναφέρονται στη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι οριζόντιο. πέρα από τα BAM και τα DCI δηλαδή. Η συζήτηση αυτή έχει ήδη γίνει σε διαφορετικό επίπεδο. Δηλαδή, ο συμβασμός για τα, μέσα, τα εξωτερικά μέσα χρηματοδότησης δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στις εσωτερικέ συζητήσεις για νέες ρυθμίσεις επιτροπολογίας. Είναι μια οριζόντια προσέγγιση που πρέπει να τηρηθεί. Γι' αυτό και είμαστε υπέρ του να μην έχουμε την οριζόντια συζήτηση εδώ στο θέμα της μπανάνας. Συνεπώ, οι υπόλοιπε αντιδράσεις μου έχουν να κάνουν με τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με τον ΠΑΜ αυτό καθ' αυτό. 1 με 6 και 8 με 10. Και έρχομαι τώρα στο τρίτο μου σημείο. Ξέρουμε ότι η συγητής υπογραμμίζει πολύ το θέμα της μείωσης της ένδυας και πρέπει με αυτόν τον τρόπο να βελτιωθεί η κατάσταση και οι συνθήκε ζωής των ανθρώπων παραγωγών μπανάνας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για ένα μέσο συνεργασία. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σχετική τροποποίηση στο DCI, που ήδη στο άρθρο 2.1 λέει ότι ο κύριος στόχος της συνεργασίας θα είναι η απάλληψη της φτώχειας στα πλαίσια της εφόρου ανάπτυξη. Είναι επίσης πολύ σωστό να μας απασχολεί η ζωή των παραγωγών μπανάνας, ιδιαίτερα των πιο μικρών, που είναι κομμάτι η παραγωγή αυτή της αλυσίδας των εσόδων. Οι προδιαγραφές ασφάλειας επίσης είναι πολύ σημαντικές. Και είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται όλα αυτά στο πρόγραμμα για την μπανάνα. Τέταρτον, βλέπω τις ειδικές τροπολογίες που προτείνονται εδώ και που πιστεύω ότι είναι πολύ επικοδομητικές. Πολλές από τις προτάσεις είναι αξιόλογες. Αλλά νομικά μιλώντας, η γλώσσα θα έπρεπε να είναι πιο συνεκτική και να συμφωνεί καλύτερα με το κείμενο το νομικό. Γι' αυτό πιστεύω ότι πολλές από τις τροπολογίες αυτές μπορούν να βελτιωθούν. Κάποιες καλύπτονται ήδη από τον DCI. Κάποιες άλλες ε, προτάσεις εδώ χρησιμοποιούν ε, γλώσσα που δεν, είναι, που δεν έχει ακρίβεια θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε αυτό με τον εισηγητή και τους συνεργάτες του και να βοηθήσουμε με κάποιες λεπτομέρειες για να βελτιωθούν αυτά τα θέματα. Πέμπτον, στην τροπολογία αριθμός 4 γίνεται μνήμα στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις ετοίμασε μία έκθεση αξιολόγησης όσον αφορά την μπανάνα. Δεν... Αυτό που μπορούμε εμείς να πούμε εδώ είναι ότι έχουμε πολλές πληροφορίες στα πλαίσια των αξιολογήσεων που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Καλό θα ήταν είτε να αποσυρθεί αυτή η τροπολογία ή αλλιώς να αναφέρονται με μεγαλύτερη σαφήνεια οι διάφορες αξιολογίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη συνέχεια, για τις χώρες που υποφελούνται από το μέσο αυτό, στην τροπολογία αριθμό 9 προτείνει ο εισηγητής να χρησιμοποιήσουμε στοιχεία των τελευταίων τριών ετών. Εδώ θέλω να τονίσω ότι Περιοριστήκαμε στα τρία διαδοχικά... Ε, δεν, δεν περιοριστήκαμε στα τρία αυτά έτη, γιατί μπορεί να μην είναι κανονικά έτη. Μην ξεχνάμε, η Τζαμάικα για παράδειγμα, ε, το 2008 περιόρισε στο μηδέν τις εξαγωγές μπανάνας, ακριβώς επειδή είχε τυφώνα. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε δίκαιοι και να μην τιμωρούμε με αυτόν τον τρόπο μια χώρα που ήδη έχει τιμωρηθεί από τη φύση μια φορά. Έρχομαι τώρα στην τροπολογία αριθμός 10. Στην τροπολογία αυτή και είπε ο εισηγητής ότι πρόκειται και για τον πυρήνα βασικά της έκθεσής του και των τροπολογιών του, εδώ απορριθμούνται διάφορα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν στις στρατηγικές στήριξης. Ίσως θα ήταν καλό να θυμηθούμε εδώ ότι προτείνονται στρατηγικές που μπορούν να έχουν διαφορετικές μορφές ανάλογα με τη χώρα. Πρώτα απ' όλα ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, δεύτερον πρόθεση της ποικιλομορφία και τρίτον ε, διεύρυνση της διαδικασίας προσαρμογής. Όλα αυτά τα στοιχεία στις τρεις αυτές περιπτώσεις, τα στοιχεία που αναφέρει η τροπολογία, εφαρμόζονται. Δεν χρειάζεται λοιπόν να γραφτούν χωριστά με την τροπολογία αυτή 10. Μια άλλη παρατήρηση για τροπολογία 10 έχει να κάνει με την εισαγωγή μιας ε, ανεξάρτητης έκθεσης. Αυτό είναι ένα συνήθιστο βήμα όταν ετοιμάζουμε στρατηγικές και είναι σαν να αφισβητούμε τις ε, ικανότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει καλές στρατηγικές στήριξης. Επίσης θα μπορούσε να οδηγήσει και σε καθυστερήσεις εφαρμογής του προγράμματος. Και έρχομαι στην τελική μου παρατήρηση, την 8η. Όπως γνωρίζετε, οι πρώτες δεσμολογικές μειώσεις για την μπανάνα γίνανε αναδρομικά 15 Δεκεμβρίου που μας πέρασε. Οι προμηθευτές μπανάνα σακέ αντιμετώπισαν την αναγκαιότητα να προσαρμοστούν, να κάνουν αλλαγές με τους χαμηλότερους δασμούς. Η ευρωπαϊκή αρρωγή είναι πολύ βασική και πήγη και πρέπει να είναι και αποτελεσματική όσο γίνεται πιο γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να δεσμευθούν ώστε να υπάρξει όσο γίνεται πιο γρήγορα μια συμφωνία. Προσδοκώ και εγώ μια καλή συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης και με τον εισηγητή κύριο Γκούρενς μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Βελγική Προεδρία έχει τώρα το λόγο που εκπροσωπεί ο κύριος Γκί Ρεγέρ. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Συμβούλιο είναι σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια πρώτη συνεργασία θα έχουμε την πέμπτη που μας έρχεται και έτσι προς το παρόν δεν έχω περισσότερες πληροφορίες να σας δώσω. Ακούσαμε και μάθαμε τι περιλαμβάνει η έκθεση βέβαια ακούγοντάς σας, αλλά θα θέλαμε περισσότερο χρόνο για να μελετήσουμε τα πράγματα. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκέρενς τώρα για να ολοκληρώσουμε την έκθεση αυτή. Παρακαλώ κύριε Γκέρενς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λέει ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όντως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και γι' αυτό και κάνουμε τις προτάσεις μας υπό μορφή τροπολογίας. Παραμένω ανοιχτός σε προτάσεις. Και εσείς και όποιος άλλος θέλει μπορεί κάλλιστα να βελτιώσει παρετέρω το κείμενό μου. Κανένας δεν έφερε αντιρρήσει σε αυτά που περιλαμβάνονται στην έκθεση από ό,τι κατάλαβα. Πάντω για την μακροπρόθεσμη στρατηγική, παρατήρηση που έγινε εξ αριστερών εδώ στην αίθουσα, λυπάμαι που δεν θυμάμαι το όνομά σα, εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Και τον έφερε και κάποιο άλλος νωρίτερα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα DCI, με ένα μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη. Μέχρι το 2013. Και αυτό γιατί υπάρχει μια λογική δημοσιονομικού προγραμματισμού που είναι αυτή που είναι και η οποία δεν φτιάχτηκε για να καταπολεμούμε την ένδια, αλλά φτιάχτηκε για να είμαστε συνεπείς και συνεκτικοί με το χρονοδιάγραμμα των διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και επίσης για να έχουμε και τα μέσα να προγραμματίζουμε τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα. Και γι' αυτό δεν μπορούμε να αναρωτηθούμε για το μετά το 2013, ακούσαμε. Εγώ όμως λέω, όχι, δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε και για μετά. Γιατί αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τους εαυτούς μας, την ανάπτυξη την θέλουμε αποτελεσματική, σωστή και διάρκειας. Η διάρκεια είναι ένα βασικό κριτήριο με το οποίο συμφώνησε όσα στην μέθοδο αξιολόγησης των προγραμμάτων, των σχεδίων και των πολιτικών αναπτυξιακής βοήθειας. Άρα, για να είμαστε συνεπείς με τους εαυτούς μας ακριβώς, πρέπει να σκεφτούμε και πέρα από το 2013. Γι' αυτό ακριβώς ζητάμε τις εξάντε αυτές αξιολογήσεις εκ των προτέρων, αλλά και ε, και μετά για να μπορούμε να διαπιστώνουμε τις ελλείψεις, τα κενά του συστήματος. Δεν αφισβητούμε τις ικανότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σίγουρα όχι της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καθ' άλλο έχω παρακολουθήσει και έχω στηρίξει με όλε μου τι δυνάμει τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μερικέ φορέ και σε αντίθεση με άλλε υπηρεσίε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε αντίθεση με ολόκληρο τον κόσμο κάποιε φορέ, γιατί συχνά είμαστε εμεί και η Εκτελεστική Επιτροπή των Βρυξελών που πρέπει να κάνουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες για να αντιταθούμε στις πιέσεις των άλλων. Μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι δεν θέλουν τίποτα άλλο εκτός από την εξαφάνισή μας. Ας αντισταθούμε λοιπόν. Γιατί αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χάνε έναν θεσμικό εταίρο ιδιαίτερα σημαντικό. Συνεπώς έχουμε κάθε συμφέρον και εσείς και εμείς να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Άρα μη θεωρείτε τις παρατηρήσεις μου εναντίον σας. Κάθε άλλο. Τώρα λέμε ότι οι χώρες παραγωγή μπανάνας πρέπει να σωματωθούν στην ανάπτυξη την περιφερειακή. Να υπάρξει ολοκλήρωση και η περιφερειακή συνεργασία. Εννοείται. Και η αξιολόγηση πρέπει να το δείξει αυτό. Τώρα υπάρχει μια ερώτηση από τον κύριο Τυρολέν για την ευελιξία. Εδώ πρέπει να ομολογήσω ότι είτε δεν πρόσεχα καλά, είτε πάντα δεν κατάλαβα ακριβώ την ερώτησή σας. Μήπως θα μπορούσατε, εφόσον συμφωνεί και η Πρόεδρο, να επαναλάβετε την ερώτησή σα, παρακαλώ. Ο κύριο Τυρολιά. Πιστεύουμε ότι για αυτό το συγκεκριμένο σημείο, όταν συγκρίνουμε τους κανονισμούς του 94 και του 99, διαπιστώνουμε ότι με τα, τους μηχανισμούς στήριξης που χρησιμοποιήθηκαν, ορισμένα βασίστηκαν στα έσοδα, το 94 αυτό, και το 99 προτιμησιακά χρηματοδοτήσαμε προγράμματα επενδύσεων. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να μπορούμε να χρηματοδοτούμε περισσότερο τα έσοδα των παραγωγών παρά να χρηματοδοτούμε προγράμματα επενδύσεων. Ή στο κάτω-κάτω να βρούμε μια ευελιξία ώστε να μπορούμε να στηρίζουμε και τα έσοδα και τα, τις επενδύσεις. Ο εισηγητής, θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μιλήσει εδώ. Έτσι όπως την εξήγησε την ευελιξία ο κύριος Τυρολιά, δεν έχει τις ίδιες βάσεις όπως κατά το παρελθόν. Ε, το δοκιμάσαμε έμεσα να στηρίξουμε τα έσοδα με διαπραγματεύσεις σε όλη τη διαδρομή της μπανάνας, έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να φροντίσουν οι παραγωγοί να έχουν περισσότερα έσοδα. Να μπορούν να παίρνουν περισσότερα. Αλλά από τη μελέτη που είδαμε διαπιστώσαμε ότι το οικονομικό προϊόν που πάει στον παραγωγό μπανάνας είναι μικρότερο κατά 2% από την τελική τιμή που τελικά πληρώνει ο καταναλωτής. Εμείς βρήκαμε ότι δεν ήταν αρκετό το ποσό αυτό. Και γι' αυτό όλο τον κλάδο της μπανάνας είπαμε ότι με άλλο τρόπο πρέπει να τον βελτιώσουμε έτσι ώστε να παίρνουν περισσότερη παραγωγή. Μένω ανοιχτό όμως τις προτάσεις σας. Αν έχετε κάποια τροπολογία ή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει κάποιο άλλο μέσο για να το πετύχουμε αυτό, είμαι ανοιχτός. Έρχομαι τώρα στην κατανομή των πόρων. Εδώ ομολογώ, παραδέχομαι, ότι δεν έχω λεπτομερέστερη πρόταση. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρησιμοποιούμε πολλά και διάφορα κριτήρια. Πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη. Θα ήθελα να είχα μία πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ξέρω ότι η Επιτροπή δεν θέλει πρόωρα να ανοίξει τα χαρτιά της, αλλά αν μη τι άλλο, εδώ, τώρα, μια που δεν παίζουμε κρυφτό, ας προσπαθήσουμε να δούμε όσο γίνεται πιο ξεκάθαρα πώς προχωράει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενημερώστε μας, σας παρακαλούμε, για τις δυνατότητες που βλέπετε εσείς σε σχέση με τα κριτήρια που εσείς έχετε επιλέξει για να βοηθήσουμε τις χώρες παραγωγούς μπανάνας. Αυτό το ονομάζει διαφάνεια ο κύριος Τυρολιά και συμφωνώ με την παρατηρήσή του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε και κάποιες ε, διαφορές σε σχέση με τις δικές μας θέσεις. Είπε ότι γενικά συμφωνούμε, τέλος πάντων αν εμείς συμφωνούμε με εσάς ή εσείς συμφωνείτε με εμάς δεν έχει σημασία αυτό, Ποιο συμφωνεί με τον προσανατολισμό ποιου, σημασία έχει να συγκλίνουν οι απόψεις μας. Εννοείται ότι όλα αυτά πρέπει να τα δούμε περισσότερο σε λεπτομέρειες. Πάντως όσον αφορά την αξιολόγηση, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και νωρίτερα. Μία ανεξάρτητη αξιολόγηση δεν σημαίνει μομφή απέναντι σε κανέναν. Και εγώ έχω υποστεί πολλές αξιολογήσεις και στο κάτω-κάτω νομίζω ότι είναι καλύτερα να μας αξιολογεί κάποιος ανεξάρτητος. Είμαστε πιο σίγουροι μετά γιατί ξέρουμε ότι έχουμε στήριξη και δεν θα μας επικρίνει κανείς. Αναφερθήκατε επίσης στα τρία χρόνια. Σε φωνώ μαζί σας. Το παράδειγμα της Τζαμάικα, στο οποίο αναφερθήκατε, είναι σωστό. Το να βασίζουμε την εκταμίευση μόνο στα τρία τελευταία χρόνια όντως μπορεί να ζημιώσει μια χώρα η οποία έχει υποστεί κάποια φυσική καταστροφή που τους έχει καταστρέψει ολόκληρη την παραγωγή μιας χρονιάς. Συμφωνώ μαζί σας εδώ να βάλουμε ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εγώ είχα βάλει τα τρία τελευταία χρόνια γιατί ορισμένες χώρες από την άλλη έχουν σταματήσει τα τελευταία χρόνια να παράγουν είτε μερικώς είτε πλήρως μπανάνα. Οπότε Καταλαβαίνετε ότι εκεί δεν πρέπει να τους δώσουμε τίποτα, γι' αυτό το έβαλε έτσι. Για την επιτροπολογία τώρα και τις κατεξουσιοδότηση πράξης, συμφωνώ απόλυτα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εδώ δεν έχω την πρόθεση να απομακρυνθώ ούτε χιλιοστό από αυτήν. Και σας το λέω ξεκάθαρα. Μην νομίζετε ότι είμαστε ξεροκέφαλοι. Μη μας βλέπετε έτσι. Μας χρειάζεστε για να περάσετε ό,τι θέλετε. Θα χρειαστείτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας στηρίξει. Οπότε καλά θα κάνετε να έχετε έναν εταίρο όπως είμαστε εμάς που θα σας στηρίξει στην καταπολέμηση και την απάλληψη της ένδυας. Μην κολλήσουμε στις συζητήσεις για τις κατεξοδότηση πράξεις. Η δικιά μας η θέση θα σας βοηθήσει τελικά. Είμαι αποφασισμένος εδώ και επιμένω. Και θέλω να είμαστε, θα έλεγα τη λέξη, συνένοχοι, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι κανένας άλλος δεν θα μας βοηθήσει όσον αφορά την ανάπτυξη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να σας το πω πιο ξεκάθαρα, καταλάβατε τι εννοώ. Πρέπει εμείς να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Αυτά ήταν τα βασικά που είχα να πω μετά από τις παρατηρήσεις που άκουσα. Επαναλαμβάνω ότι είμαι ανοιχτός. Και εγώ και οι συνεργάτες μου που με βοήθησαν να εκπονήσω το κείμενο αυτό. Ό,τι προτάσεις έχετε εσείς, οι συνάδελφοι δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είμαι στη διάθεσή σας. Και ελπίζω να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας όσο γίνεται πιο γρήγορα. Όσον αφορά τώρα το οριζόντιο διάβημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είπα ότι είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας. Ευχαριστούμε. Να σας υπενθυμίσω για τις τροπολογίες. 15 Σεπτεμβρίου στις 6 λίγη προθεσμία. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στην επόμενη συνεδρίαση 4 και 5 Οκτωβρίου. Θα προχωρήσουμε τώρα στις ψηφοφορίες που προβλέπονταν για τις 4.30 και το σημείο 10 της ημερής διάταξης, ο Δημοκρατικός Έλεγχος του Προγραμματισμού στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την ανάπτυξη. Θα επανέλθουμε μετά από τις ψηφοφορίες. Σας καλώ λοιπόν να βγάλετε τις κάρτες ψηφοφορίας. <clears throat> nous allons voter sur la modification du règlement. Θα ψηφίσουμε για την τροποποίηση του κανονισμού 1605 του 2002 που αφορά την θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο Γενικό Προπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Έχουμε λοιπόν το άρθρο 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε για το σύνολο της πρότασης όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Euh, la possession du Parlement sur le projet du budget tel que modifié par le Conseil. Τώρα, η θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο. Euh, Για το προπολογισμό λοιπόν θα ψηφίσουμε unblock. Υπάρχουν τέσσερα μπλοκ. Πρώτο. Περιλαμβάνει πέντε τροπολογίες. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Non, c'est, vote pour moi. Voilà. Donc le vote est ouvert. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Δεύτερο σύνολο τροπολογιών. Δύο τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Tout le monde a voté. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνονται. Τρίτη ομάδα τροπολογιών, ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τώρα, περνάμε στο τέταρτο σύνολο τροπολογιών που αποτελείται από τέσσερις τροπολογίες. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. Τώρα ψηφίζουμε μία προς μία τις υπόλοιπες τροπολογίες. Η τροπολογία 5407, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. 54-15 καταπίπτει και αντικαθίσταται από την προφορική τροπολογία που φέρει τον αριθμό 54-32. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54-0. Ψηφίζουμε. Ψηφίζατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54.01. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 02 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 5406. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-19. Ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-20. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-21. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-22. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-33 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-24. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-25. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-26. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-27. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Πέντε Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54-29. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 5,430 54-30. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τελειώσαμε. Λοιπόν, για τον προϋπολογισμό λοιπόν τελειώσαμε. Όλες οι τροπολογίες εγκρίθηκαν. Τώρα θα ψηφίσουμε για την έκθεση της Βερονίκη Ντεκεζέρ.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 Λοιπόν, προχωράμε στη ψηφοφορία τη έκθεση τη κυρία Βερονίκτη Τικιζέρε. τροπολογία 10. Ψηφίζουμε. Τέλο τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλο ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 12. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 13. Τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16. Ψηφίζουμε για το 16. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. πέρα τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20. Άργεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 22 καταπίπτει. Πάμε στην 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 25. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 26. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 27. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 29. Είναι προφορική τροπολογία της κυρίας Στόγια, που θα μας την παρουσιάσει κιόλα. Ναι, δέχομαι. προφορική τροπολογία στην 29 της κυρίας Τόγια. Η τροπολογία έχει ως εξή. Λέει ότι δεδομένου στη σημαντικού ρόλου που παίζει για στην πρόθεση της εκπαίδευσης της δημόσιας υγείας, οι μη κρατικές ε, οργανώσεις συμπεριλαμβανομένων των θρησκευτικών οργανώσεων στα ιδιωτικά ε, νοσοκομεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Including που λέει εκεί. Including. Αυτός είναι ο όρος που προστίθεται. Μάλιστα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ο ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30. Τροπολογία 30 ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Ζητείτε χωριστή ψηφοφορία. Η κυρία Τικεζέρ θέλει να το σχολιάσει. Όχι. Ωραία, χωριστή ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το πρώτο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 34. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 35. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Έγκρινεται. Τροπολογία 37. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 38. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39, άρχεται ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Τροπολογία 40, άρχεται ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 41, ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 42, Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 43. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 44. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 45. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 47. Απορρίπτεται. 48. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 49. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 50. Άρχεται την ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 51. Ανοίγει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Ανταπτή. Εγκρίνεται. Τροπολογία 52. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 53 ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 54 ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 55 άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 56 ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορία. ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 57. Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία. εγκρίνεται. 58. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 59. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι, τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 60. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. το. 61. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 62. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 63. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 64. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 65. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 66. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 67. Άρχεται ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε για, για τα εκτιμώντας. Συμφωνείτε να τα ψηφίσουμε on Όχι. Ωραία λοιπόν. Είναι μπερδεμένο. Α τα ψηφίσουμε ένα-ένα. Τέσσερα. Ψηφίζουμε για το τέσσερα. Τέλο ε, τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τρία. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τα υπόλοιπα unblock. Λοιπόν, unblock ψηφίζουμε από το 5 μέχρι το 9. Υπέ, ε, ψηφίζουμε Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εγκρίνονται. On vote sur les Λογικές σκέψεις. 1. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορία ε- Εγκρίνεται. Και 2. Ψηφίζουμε, ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Ψηφίζουμε τώρα για το κείμενο ολόκληρο της έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Θα ψηφίσουμε τώρα. Το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, σχετικά με τη διάσκεψη του Κανκούν. Τροπολογία 6 καταρχήν. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. 7. Άρχεται ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 9. Ο κύριος Γκερέρο. Στα ισπανικά, στα ισπανικά λέω, η τροπολογία αυτή στις τελευταίες γραμμές λέει ότι δεν έχει προχωρήσει αρκετά το θέμα ε, των, της ανάπτυξης, ενώ πρέπει να μιλάει για το περιβάλλον εδώ στην πολιτική συνεργασίας και ανάπτυξης. Εδώ πρέπει να γίνει μια διόρθωση γιατί δεν είναι σωστό το ισπανικό κείμενο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Θα λάβουμε υπόψη μας βέβαια την παρατήρησή σας. Ψηφίζουμε τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 11. Άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Άρχιδη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας. Α, δεν λειτουργεί. Για να ξαναρχίσουμε την ψηφοφορία, γιατί κάποια μηχανήματα δεν λειτουργήσαν. Λοιπόν, άρχισε η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Άρχισε η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Συγγνώμη. Τροπολογία 15 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχισε ψηφορία για το πρώτο τμήμα της 15. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 16. Έχει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. έχει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 18. έχει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπόλη 19. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τι έχουμε άρχη ψηφοφορία. 2. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Άρχιτη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Άρχιτε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας Δεν λειτουργήσε το σύστημα. Να ξαναρχίσουμε. Τροπολογία 5 πρώτο τμήμα. Άχι ψηφοφορία. Λειτουργεί τώρα. Ε, θα προσθέσουμε τη δική σας ψήφο. Ça marche. D'accord. <laughs> Le vote est clos. Ωραία, λειτουργεί τώρα. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα τη 5. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Καναφορά φορά τροπολογία 1. Άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας πληροφορίες. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία. Ένα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται το σύνολο του κειμένου ως τροποποιήθηκε. η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Nous Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες και μπορούμε να επανέλθουμε στο σημείο που κατά βάση έπρεπε να έχουμε εξετάσει πριν την ψηφοφορία. Σημείο 10. δημοκρατικό έλεγχο του προγραμματισμού στο πλαίσιο τη νομοθεσία για την ανάπτυξη. Και πρέπει τώρα να προχωρήσουμε στον δημοκρατικό έλεγχο των εγγράφων προγραμματισμού, ενδεικτικά προγράμματα εθνικά και περιφερειακά για τη Βραζιλία, το Μερκοσούρ και την ε, κοινότητα των Άνδεων. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκέρενς, που είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας ΔΕΛΤΑ, για να μας παρουσιάσει τις, ε, τα συμπεράσματα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Δεν θα αναφερθώ από τις ουσίες. Θα την μονάχα μία τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος και θα ήθελα να προβλέψουμε πρώτα μία συζήτηση μεταξύ των συντονιστών για το θέμα αυτό. Συμφωνούν όλοι, ρωτάει η Πρόεδρος, να εξετάσουμε το θέμα καταρχήν μεταξύ των συγητών. Ο κ. Γκερέρο. Ναι, δεν διαφωνώ να δουν οι συντονιστές αυτό το σημείο. Αναρωτιέμαι όμως τελικά μετά τη συνεδρίαση των συντονιστών δεν θα πάει στην ομάδα εργασίας Δέλτα. Οπότε επαφίομαι στον κύριο Γκούρενς. Ό,τι εκείνος αποφασίσει, εντάξει. Να το δουν οι συντονιστές και μετά η ομάδα Δέλτα ή να το δει κατευθείαν η ομάδα Δέλτα. Ό,τι εκείνος προτιμάει. Επαφίομαι σε αυτόν. Κύριε Γκρέσ, θα ήθελα να υποστηρίξω αυτά που είπε ο κ. Γκερέρο. Φαντάζομαι να μην διαφωνεί κανένα να συζητήσουμε πρώτα μεταξύ των αυτό το θέμα. Έτσι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα σημασία, στα διάφορα δηλαδή. Δεν έχει ζητήσει κανένα να εγγραφεί τίποτα στη διάφορα. Οπότε, α, ο κύριος Γκέρεντς. Μπορούμε να προβλέψουμε τις συνεδρίες των συντονιστών αμέσως μετά το πέρα της μας. Αν οι άλλοι συμφωνούν, θα μπορέσουμε να κερδίσουμε πολύ χρόνο. Να μην περιμένουμε δηλαδή μέχρι έξι 6, να συνεχίσουμε αμέσως. Πρώτα συμφωνούν οι συντονιστές. Ωραία. Να, προ... να ειδοποιήσουμε τον κύριο Μίτσελ μόνο. reste plus que les dates des prochaines réunions. Donc c'est à Bruxelles. δεν σας είπα πότε θα είναι η επόμενη μας συνέντευξη. Αύριο στις Βρυξέλλες εδώ, 3η, 31 Οκτωβρίου. 2 με 3,5, μια έκτακτη συνέντευξη για το Πακιστάν. Σας καλώ όλους να έρθετε να ακούσετε την κυρία Γεωργίευα.